Colleagues, can I bring the meeting to order and remind you, I think... Μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι θα περάσει στην αυτόματη αναμετάβαση web stream. Έχετε τη μεσαία διάταξη μπροστά σας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτή. Σας ευχαριστώ. Έχετε και τα πρακτικά της 28 Φεβρουαρίου. Συμφωνούμε και πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ. To number three, can I just introduce to... Περνάμε στο σημείο 3. Ο ε, Πρωθυπουργό θα δείτε ότι είναι παρόν εδώ και χαιρετίζουμε στη συνεδρία τη Επιτροπή Μεταφορών. Επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη. Next item on the agenda is the action plan on. Το επόμενο είναι το πρόγραμμα δράση για τα παγκόσμια συστήματα πλοϊκή μέσω δεζιφορού μεταφορέ. Η κυρία Τίκα είναι η συγκεκριά μα. Președinte, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους συναδέλφους που μου συνεργάστηκαν, ιδίως και εδώ στους με τους οποίους συνεργαστήκα πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι το θέμα αυτό που σχετίζεται με το παγκόσμιο σύστημα υπολογίσης μεσοδορυφόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό σύστημα. Γι' αυτό, πλιστάκης, ζήτησα και μέσα στο πολιετές αυτό πρόγραμμα χρηματοδότηση να υπάρχουν πόροι για ε, έρευνα στους διάφορους τομείς εφαρμογής του συστήματος. Το ίδιο θα ισχύσει και για το την επόμενη χρηματοδοτική και προγραμματική περίοδο. Και εκεί έχω ζητήσει να υπάρχουν είπα για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τα συστήματα Γαλιλαίο. Όλα τα άλλα συστήματα έγνωση κλπ. θα αντικαταστοστούν από το σύστημα Γαλιλαίο όταν έχει ετοιμαστεί αυτό. Είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό για τη μελλοντική εφαρμογή και την εκμετάλλευση του δυναμικού να υπάρχουν ήδη τώρα επενδύσεις σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τομέα των μεταφορών. για την αστική προστασία, για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές και γι' αυτό θεωρώ ότι πρόκειται για ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή του τις απαραίτητες, τους απαραίτητους πρόπους. Έχουμε 48 τροπολογίες. Καταρχήν δεν υπάρχουν προβλήματα με τις τροπολογίες αυτές. Προσπάθησα να λάβω υπόψη τις απόψεις των συναδέλφων. Νομίζω το καταλήξαμε σε καλούς συμβιβασμούς και ενδιαφέρομαι να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να μην με ακριβωρήσω περαιτέρω, απλώς να τονίσω και για μια φορά πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι χρειάζεται για τον καθορισμό των προτεραιότητων στο επόμενο πολιετές πρόγραμμα χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, από στρατηγικής απόψεως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για μια προσπάθεια που έχει γίνει από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το σύστημα Galileo, το οποίο υπάρχει και λειτουργεί, το GNSS είναι ένα σύστημα που σαφώς έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν προγράμματα και αυτό που είναι σημαντικό είναι τα πρότυπα και βεβαίως η χρηματοδότηση που γίνεται μέσω του προγράμματος Γαλιλαίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και όλα αυτά βεβαίως συνδέονται με την χρηματοδότηση. Το θέμα της ασφάλειας ε, όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές. Θέματα πολύ σημαντικά. Επίσης θέματα που έχουν σχέση με τις χερσαίες μεταφορές, με τους σιδηροδρόμους. Όλα αυτά τα οποία βεβαίως μπορεί να ρυθμιστούν με ένα τέτοιο σύστημα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, η οποία πραγματικά μπόρεσε, βάσει των πολλών τροπολογιών που είχαν υποβληθεί, να δημιουργήσει τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα συστήματα πλοήγησης που υπάρχουν και λειτουργούν. Το GPS, αλλά υπάρχει και το σύστημα το κινέζικο. Θα πρέπει να υπάρξει συμβατότητα, ναι, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε από κοινού. Επίσης, σήμερα που βλέπουμε την καταστροφική δράση που μπορεί να έχει η φύση στον πλανήτη μας. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι σήμερα πολύ σημαντικά. Η γεωγραφική χρησιμοποίηση όλων αυτών των ε, προτύπων. Σήμερα βλέπουμε οι περισσότερες τροπολογίες των συναδέλφων να μας οδηγούν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη να καλυφθεί η νοτιοανατολική Ευρώπη, η Βόρεια Αφρική, η αποτελεσματικότητα επίσης αυτών των συστημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το θέμα του κόστους και βεβαίως αυτό που μας αφορά εδώ ιδιαίτερα είναι να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης. Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων επηρεάζει άμεσα, βεβαίως, επηρεάζεται άμεσα από τα ποσά που διαθέτουμε. Σε δύο χρόνια θέλουμε να αρχίσει να λειτουργεί 100% το σύστημα Γαλιλαίο και τα συστήματα υλοποίησης δεν μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Ο κύριος Δουρικέ έκανε μια πολύ σωστή πρόταση μέσω της τροπολογίας τους και όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε κάποια από τα αποτελέσματα αυτού του συστήματος να μπουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα θέλαμε να υποβάλουμε και δύο προφορικές τροπολογίες από μέρους της, ε, του ΕΛΚ. Στην ε, παράγραφο 11, συμβαστική τροπολογία 2, να προσθέσουμε εδώ, μεταξύ των λέξεων GNSS, και Enable Transport να βάλουμε εδώ μία αναφορά, μία φράση που να αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Σας το προτείνω προφορικά και ιδιαίτερα μία άλλη τροπολογία, μία άλλη αλλαγή στην παράγραφο 3 Ζητάει από την Επιτροπή να διασφαλίσει για το σύστημα έγνος, για την πολιτική αεροπολία, για τις αρμόδιες αρχές ή μέσω των αρμοδίων αρχών και εδώ να βάλουμε μια τελεία και να σβήσουμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά την εισηγήτρια και όλους τους συναδέλφους που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το αποτέλεσμα. Sorry, I think my microphone went off. Mrs. Jensen. <laughs> Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τικάο γιατί ε, είδα με θετικό μάτι και τις δικές μου τροπολογίες και τις τροπολογίες ομάδας Άλντε και τις συμπεριέλαβε σε σχέση με το ITS και άλλα ζητήματα. Υποστηρίζω τη θέση της εισηγήτριας Στηρίζω και τις ε, συμβιβαστικέ τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν. Δεν ήμουν βέβαια απολύτω, βέβαιη για το όλο αυτό ζήτημα ε, της επέκτασης και της ε, στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Αλλά τέλος πάντων αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την άποψή σας. Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστό, έτσι θα πράξουμε και εμείς λοιπόν κυρία η Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να είναι εφικτό. Να φροντίσουμε να είμαστε βέβαια ότι μπορεί να είναι εφικτό. Μεταξύ των θετικών χαίρομαι επίσης που έγινε δεκτή η τροπολογία κόσα για την προσβασιμότητα που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αναφερθεί. Επίσης ε, δεν ήμουν βέβαιη για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο κύριος Κούν έκανε μια σχετική αναφορά Πράγματι έχουμε διαφορετική τεχνολογία γι' αυτό, αλλά νομίζω σωστά τα είπατε. Θα πρέπει και στον τομέα αυτό να κάνουμε έρευνα στο σχέδιο δράσης και να δούμε πώς το GNSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, για σκοπούς των θαλάσσιων μεταφορών. Και πράγματι, μία από τις ιδέες που είχαμε ήταν ότι οι εφαρμογές του Γκαλιλαίου θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές ε, με άλλες τεχνολογίες. Δηλαδή, αν δούμε ότι πράγματι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυτό θα το εκτιμήσει η αγορά ε, και για το μέλλον και θα έχουν πλεονέκτημα, θα έχουν προτεραιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τικάου για την πολύ καλή δουλειά της. Ευχαριστώ. Λίχτεμπεργκερ για τους πρασίνους. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Τι να πω ότι τον ληφθεί υπόψη αυτό που είπε ο κύριο Κούν για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Μου φαίνεται πάρα πολύ λόγο που θα το υποστηρίξω. Επίξω στο θέμα της διαλειτουργικότητας που είναι τόσο έντονο στην εκθεσεφή μου φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό. Γιατί αυτά τα συστήματα θα μπορούν να ωφελήσουν ιδιαίτερα και να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα μόνο αν είναι διαλειτουργικά και ευρέως εφαρμόσιμα όταν προσπαθήσαμε παλαιότερα να υποχρεωθούν όλοι με ένα σύστημα και μοναδικό να αγοράσουν νέε συσκευέ, δεν μου φαίνεται ότι είναι κάτι που θα μας βοηθήσει για το μέλλον. Και γι' αυτό το θέμα της γενετοικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω προβλήματα με κάποιες τροπολογίες που αφορούν χρηματοδότηση. Γιατί το οι συνήθεις άγουσα δηλαδή να κοινωνικοποιηθούν ε, τα κόστη και όχι και τα κέρδη, μου φαίνεται ότι είναι πολύ προβληματικό. Έχω λοιπόν το πρόβλημα ότι προφανώς ε, δεν μπορέσαμε να εντάξουμε μία πάρα πολύ σμάδα λίτου ε, χρηστών, εκείνο δηλαδή που θα έρθουν αργότερα, Äh, Γιατί θα πρέπει να δούμε ποιος ενδιαφέρεται και ποιος χρησιμοποιεί και ποιος εργάζεται πάνω στα συστήματα αυτά. Και γι' αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω με εσάς από τις τροπολογίες. Γιατί εποχές όπου ο, ο δημόσιος κορβανάς είναι σχετικά ισχνός και άδειος, θα πρέπει να ε, βρούμε μια άλλη λύση που να υπάρχει συμμετοχή όσον αφορά το κόστος και όσον αφορά το κέρδος. Να μην έχουμε λοιπόν μια άδικη κατανομή. για να μπορέσουμε στο μέλλον να παίξει το σύστημα αυτό ένα σημαντικό ρόλο διεθνώς και παγκοσμίως. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Τίκα. Νομίζω ότι πολλές από τις τροπολογίες είναι εντάξει, είναι αλληλοσυμπληρούμενες σε ό,τι αφορά την έκθεση της κυρίας ε, Τικάου και συμπληρώνω και την έκθεση εν γέννη. Έχω δύο σχόλια να κάνω σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Γέννησεν μόλις πριν, δηλαδή Μπορεί να μην είναι δορυφορική πλοήγηση ε, το κατάλληλο, η κατάλληλη τεχνολογία, γιατί υπάρχουν άλλες τεχνολογίες που μπορεί να λειτουργούν σε κάποιους τομείς και είναι σωστό. Αυτό πρέπει να κάνουμε έτσι μια σύγκριση ε, του ποια τεχνολογία είναι καλύτερη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, στη 34 τροπολογία λέγεται καλείται η Κομισιόν να δει κατά πόσον τα έσοδα από δραστηριότητες σχετικές με το Γαλλίο θα μπορούσαν να ε, πάνε στον προπολογισμό. Τι θα πει αυτό ακριβώς, θα μπορούσε να σημαίνει χίλια πράγματα. Πού θα πάνε, σε ποιο ακριβώς ε, κονδύλιο αναφερόμαστε. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από χρήματα των φορολογουμένων. Αν δει κανεί όλο το επιπλέον κόστος ε, που θα πρέπει να έχουμε για την έρευνα, την τεχνολογία, την επιτεύξη προόδου, εγώ θα ήθελα να έχουμε ε, κάποιε διευκρινήσει σε ό,τι αφορά την Τροπολία 34 ΡΙΚΕ. Πού θα μπορούσαν να χωρούνται στο προπολογισμό. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί, τέλος πάντων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών, είπα είναι εντάξει, αλλά έχουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Είτε μας αρέσει είτε όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι θα γίνει ακριβώς. Τελικά ε, το Γαλιλαίο ε, χρηματοδοτήθηκε από δημόσια κονδύλια γιατί ο ιδιωτικό τομέα δεν χρηματοδότησε επαρκώ. Πρέπει να το δούμε αυτό. Επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ω προ το σημείο αυτό. Και κάτι τελευταίο. Έχουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα μπορούσε να μας κάνει μια ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με το σχέδιο δράσης, πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί φυσικά εδώ εμείς μπορούμε να τα συζητάμε όλα αυτά, αλλά καλό θα ήταν να μας δώσουν και μια γενική επισκόπηση από πλευράς κομισιών. Και τώρα θα πω το τελευταίο. Εντάξει, μπορούμε να περιμένουμε ίσως, αλλά σε ό,τι αφορά την τροπολογία 10 έχουμε ένα ερωτηματικό για την πλήρη ικανότητα ανάπτυξης του συστήματος Γαλιλαίου. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Το σύστημα Γαλιλαίο θα αναπτυχθεί στην πλήρη ικανότητά του. Και ένα τελευταίο για τη Βόρεια Αφρική και κάποιες άλλες περιοχές. Και πάλι δεν είμαι απολύτως βέβαιη σε σχέση με τη λήψη της σχετικής απόφασης, αν δει κανείς τις αρχικές συζητήσεις που είχαμε με τον, για τον Γαλιλαίο και για την προσχώρηση τρίτων χωρών, είναι για πολιτικό το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσον λοιπόν είναι σκόπιμο τώρα στο Συμβαστική Ένα να, ε, να έχουμε αυτή τη διατύπωση. Ε, δεν είμαι πεπισμένη για τη συμπερίληψη των χώρων αυτό. Πάντως, την ισχύτρια θέλω να την ευχαριστήσω και φυσικά θα ακούσω και τα σχόλια των υπόλοιπων συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τικάου για την ε, ποιοτική δουλειά της που καταλήγει σε μια ευρεία συνένεση. Το σύνολο του προβλήματος είναι οικονομικό, θέλω να τονίσω. Όλοι συμφωνούν με τη σημασία επί της αρχής, ε, τη σημασία του συστήματος, την ανάπτυξη του. Ενδιαφέρει επίσης ε, πάρα πολλά θέματα των μεταφορών, την διαλειτουργικότητα, από τη διαλειτουργικότητα μέχρι την ασφάλεια. Αλλά το πρώτο, όπως είπε και ένας συνάδελφος, είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε ο ιδιωτικός τομέας να κάνει επενδύσεις. Είναι πολύ διάζουσα κατάσταση. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα τέτοιου τύπου όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτού του προγράμματος. Ε, πρώτο πρόγραμμα λοιπόν είναι το οικονομικό. Υπάρχει έλλειμμα στις επενδύσεις, δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις. Λείπουν περίπου δύο δις και δεν ξέρω πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά. Υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα που αναφέρω και στην τροπολογία 35 ε, και εδώ επανέρχομαι στην παρατήρηση της κυρίας Φώστερ ε, για την 34. Έχουμε για τη διάχυση τήρηση του συστήματος, για τη συντήρηση του συστήματος ε, πρέπει να δαπανηθούν 800 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, αν υπάρχουν έσοδα από την εκμετάλλευση, τουλάχιστον θα πρέπει να δοθούν στον υπεύθυνο, στην Κομισιόν, για να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον εν μέρη αυτά τα έξοδα ε, συντήρησης. Το... Και δεν νομίζω ότι τα έσοδα θα είναι επαρκή για να καλύψουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπε και μια συνάδελφος, ο ιδιωτικός τομέας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε επενδύσεις. Επομένως, δεν θα ήθελε να... Δεν θα ήταν σωστό μάλλον να ενταχθεί τώρα στο σύστημα και να υποφεληθεί από την ε, θέση σε εμπορία. Επίσης, η ανάπτυξη των ε, εφαρμογών θα πρέπει να είναι υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση. Ε, τροπολογία τροπολογία 34 και 35 πάνε, πρέπει να τις δούμε από κοινού. Θα υπάρξουν έσοδα από την εκμετάλλευση του συστήματος, τουλάχιστον για το hard. Το 34 ζητάει αυτά τα έσοδα να πάνε στην Ευρώπη και επομένως έτσι ε, ρυθμίζουμε εν μέρη το πρόβλημα που θέτει η τροπολογία 35, δηλαδή πώς θα βρεθούν αυτά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Συνδέονται λοιπόν οι τροπολογίες 34 και 35. Τελειώνω λοιπόν. Όλοι συμφωνούν, κανένας δεν ξέρει πώς θα πληρώσουμε για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και τελικά πώς θα λειτουργήσει και πώς θα το πληρώ. Πού θα βρούμε δηλαδή τα λεφτά για να λειτουργήσει, τα λειτουργικά έξοδα. Μιλάω δηλαδή για τις δύο τροπολογίες που συνδέονται και όλες 34 και 35. Δύο σύντομα σχόλια. Συμφωνώ με την παρατήση Φώστερ για τις εφαρμογές, τη διεύρυνση των εφαρμογών του συστήματος. Δεν θυμάμαι πότε, αλλά υπήρχε μία έκθεση από μία ομάδα επιστημόνων, νομίζω, που προειδοποίησε ε, για αυτό το τεχνολογικό ε, μπέρδεμα. Όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα, Πρόεδρε, θυμάστε ότι ένα από τα προβλήματα που είχα εντοπίσει ότι δεν υπάρχει ε, του συστήματος εναντίον του ηλεκτρομαγνητικού παλμού ή παλμών. Ε, αυτοί οι επιστήμονες από την Οξφόρδη προειδοποίησαν ότι μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο ένα τμήμα του ας πούμε, θα ελέγχει ας πούμε, όχι μόνο τις ενέργειες μεταφορές αλλά και τις θαλάσσιες μεταφορές, τότε μπορεί ε, να καταρρεύσει όλο μαζί. Ε, γι' αυτό προσοχή. Δεν έχει νόημα να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την ε, τεχνολογία ε, σε διάφορα είδη μεταφορών. Δεύτερο, δεύτερο σχόλιο, το οποίο έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι για τη χρηματοδότηση. Άκουσα αυτό που είπε ο κ. Ρικέ, για το, τα ποσά που χρειάζονται, ιδίως για τη συντήρηση του προγράμματος αυτού. Αλλά και κάτι που είχε πει ξεκάθαρα η Επιτροπή μας στο παρελθόν είναι ότι η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει τη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων TENS. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, δηλαδή, ότι έχουμε και άλλα χερσαία προγράμματα, τα οποία θα πρέπει εν μέρει να χρηματοδοτηθούν ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρότι αυτό είναι εμβληματικό πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε αποκλείοντας ε, άλλους, άλλες χρηματοδοτήσεις. Θα ήθελα να το θέσω λοιπόν αυτό για να μην χρηματοδοτήσουμε λοιπόν το σύστημα αυτό Γαλιλαίος εις βάρος άλλων συστημάτων, εις βάρος άλλων προγραμμάτων TEN. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα ε, για μια τροπολογία συγκεκριμένη, της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την παρακολούθηση, Τι σκέφτεται ακριβώς κυρία Σέντερ ε, όταν λέει για ασφάλεια, μιλάει για safety security, γιατί στα αγγλικά οι δύο όροι είναι διαφορετική και έχουμε και θέματα απορρίτου των δεδομένων. Άρα, τι ακριβώς εννοεί η κυρία Αγιάλα. Γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί και το αν θα δεχθώ ή όχι την τροπολογία, διότι τι εννοούμε ασφάλεια παρακολούθηση. Safety ή security. It is safety. Safety, safety είναι στα αγγλικά το νόημα. Ε, αυτό ήθελα να πω. Την ασφάλεια ε, υπό αυτή την έννοια, οδική ασφάλεια κτλ. Και τις εμπορευματικές μεταφορές, την αλασιμότητα των εμπορευμάτων. Συνήθως έχουμε πρόβλημα στον τομέα αυτό. Μιλάω για αυτή την πλατφόρμα υπηρεσιών για τον πολίτη. Δεν μιλάμε για στρατιωτική ασφάλεια και τέτοιου είδους πράγματα. Ε, ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος. Safety στα αγγλικά λοιπόν. Ο κύριος Στίγμαν από την Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Τικάου για την εξαιρετική της έκθεση. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικά τα όσα περιέλαβε στην έκθεσή της και σε σχέση και με την αρχική πρόταση της Κομισιόν νομίζω ότι προσθέτει αξία. Σε ό,τι αφορά την αξία του Έγνος και του Γκαλιλαίου για τον τομέα των μεταφορών, νομίζω ότι έχουν υποθεί πολλά. Είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο για τον τομέα των μεταφορών κατά την άποψη της Κομισιόν. Και για τα ευρωπαϊκά δίκτυα να πω ότι το Γαλιλαίο και το Έγνος είναι εξέχουσα σημασία στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων γιατί θα δώσουν ένα είδος ευφυΐας, αν θέλετε, ε, σε αυτή την ε, όλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις υποδομές και εμέσως θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πόρων με πιο ευφυείς συναλλαγές και θα ε, βελτιωθούν επίσης και τα περί ασφαλείας, οι διατάξεις ασφαλείας. Θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις σε τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει πολύ μεγάλη ε, σχεση κόστου κόστους-οφέλους, πολύ θετική αναλογία και να πω και μια κουβέντα για τις τροπολογίες. Νομίζω ότι οι περισσότερες τροπολογίες είναι ευπρόσδεκτες από πλευράς κομισιών Αυτό το οποίο αφορά την περιφερειακή συγγνώμη, κάλυψη που επισημάθηκε από αρκετού ομιλητέ. Θέλω να σα πω ότι για εμά η κάλυψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όλα τα άλλα έπονται. Βέβαια, μας ενδιαφέρει, επειδή ακριβώς βλέπετε ε, το όλο ε, σύστημα και την κάλυψη, καλύπτεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η Μέση Ανατολή από το ΟΒΕΤ και το βόρειο τμήμα της Αφρικής και το σύνολο της Αφρικής. Εμείς προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη διεύρυνση, την επέκταση του πεδίου εφαρμογή, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το δευτερεύον. Το υπαριθμό 1 είναι η πλήρης ευρωπαϊκή κάλυψη. Και να πω και δύο-τρία πράγματα για τη χρηματοδότηση και για την διάμεση αξιολόγηση, γιατί τέθησαν κάποια πολύ σημαντικά ε, πράγματα. Κατά το παρελθόν και υπό τις παρούσες δημοσιονομικές προπτικές έχουν υποχρεωθεί 400 και περίπου εκατομμύρια από τους πόρους των εφαρμογών που προβλέπονταν να τα χωρίσουμε για την οικοδόμηση αυτού του όλου συστήματος. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά μεταφέραμε κάποια χρήματα από τις εφαρμογέ προς τις υποδομές και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα των εφαρμογών γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τη βιομηχανία μας και σε ό,τι αφορά τα έμεσα ωφέλη, τα χρήματα, το χρήμα πραγματικά βρίσκεται στις εφαρμογές. Μιλάμε για δις, για δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Και όσο καλύτερα ε, καταφέρουμε να τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό όλη την αγορά την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία, καλύτερη, τόσο καλύτερο θα είναι και η απόδοση που θα έχουμε από τι επενδύσει αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τικάου, να προσθέσετε κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και όλους εκείνους τους αδέλφους που ζήτησαν το λόγο και επίσης να ευχαριστώ την Κομισιόν για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε συμπληρωματικά. Και θα ήθελα να προσθέσω ένα σημείο. Είναι πάρα πολύ σημα... μεγάλη στατική σημασία στο πρόγραμμα αυτό και το έγνος επίσης και το ελαίος θα πρέπει να... να τονίσουμε ότι αυτά τα συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πολιτική χρήση και θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε και συμβατά με το σύστημα GPS. Και όταν εφαρμογηθεί πλήρω το Γαλιλαίο θα έχουμε καλύτερη κάλυψη, μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή και ισχυρή εφαρμογή και στις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπαν διάφοροι από τους συναδέλφους. Ελέγχθη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το πλήρες σύστημα. Έχουμε το έγνος τώρα, αλλά για να μπορέσουμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται, είναι σημαντικό να φροντίσουμε την εφαρμογή του ζητήματος Γαλιλαίου. Να μην σταματήσει δηλαδή εν μέση οδό, θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως για να μπορέσουμε να έχουμε και το μέγιστο όφελος. Ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω το ξεκίνητα για τι δικαίωση, είπε και το είπε και η Κομισιόν, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βέβαια η κάλυψη όλης της ευρωπαϊκής επικράτειας. Και κατά δεύτερο λόγο μπορούν να σκεφτούν κάλυψη και άλλων περιφερειών. Η κύρια προτεραιότητα είδα η κάλυψη όλης της επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις Τη κύρια Λίχτεμπεργκερ και του κυρίου Μπρέτμαν όσον αφορά το χρηματοδότηση και η κυρία Φώστορ αναφέρθηκε μάλιστα στο ίδιο σημείο. Θα ήθελα να πω αυτό που η αναφέρει στις τραπολογίες του κύριου Ρικέ που θα ήθελα και να υποστηρίξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι πόροι όχι μόνο για την ανάπτυξη τη απαραίτητη υποδομή για τους δορυφόρους και όχι μόνο για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε, αλλά είναι ταυτόχρονα σημαντικό κατόπιν να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για την ε, ε διαχείριση ετήσια. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι εν λόγω τροπολογία του κυρίου Ρικέ εξετάστηκε προσεκτικά από μένα σε σχέση και με αυτά που είδαμε στο παρελθόν. στην ε, περασμένη θητεία είχε μπλοκαριστεί το θέμα γιατί στην αρχή πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από μια ιδιωτική και δημόσια σύμπραξη, πράγμα που δεν ήταν δυνατόν τελικά, γιατί τελικά εφόσον πρόκειται για ένα δημόσιο σύστημα θα πρέπει να διαθέσουμε και δημόσιους πόρους που θα αναφέρονται στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα Γαλιλαίο συγκεκριμένα και μου φαίνεται γι' αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για πώς στηρίζω αυτές τις τροπολογίες καθώς και την τροπολογία της κυρίας Γέντζεν. Χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση για τον Γαλιλαίο και για το έγνος. Ε, ταυτόχρονα όμως δεν θα ήθελα αυτοί οι απαραίτητοι πόροι να αφαιρεθούν από άλλα σημαντικά προγράμματα υποδομής. Και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα και με την τροπολογία της κυρίας Γέντζεν. Θα ήθελα να τονίσω ότι ανάφερα με την ε, μεσοπρόθεσμη, ε, ταυτόχρονα με την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση να δούμε πού θα χρησιμοποιηθεί μέχρι τότε το θέμα. Αυτά κύριε Πρόεδρε θα, θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλου του συναδέλφου, Καθώ επίση και την Εκτελεστική Επιτροπή και ελπίζω να ευχαριστώ. That Ωραία. Ολοκληρώνουμε την εξετασία του θέματος στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο είναι οι διεθνεί ε, συμφωνίε αεροπορικών μεταφορών μέσα στα πλαίσια τη συνθήκης της Λισαβόνας, η δική μου έκθεση δηλαδή. Υπήρξαν 15 τροπολογίε για το σχέδιο αυτό έκθεση και μπορώ να συμφωνήσω με 12 εξ αυτών. Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια προφορική τροπολογία. Θα μπορούσα και με αυτή να συμφωνήσω. Πολλέ από τι τροπολογίε αυτέ θεωρώ ότι κινούνται προ σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να σα επενθυμίσω ότι αυτή είναι μια έκθεση που ίσω έχω να ορίσει ένα πλαίσιο. Δεν είναι μια έκθεση που υπησέρχεται σε όλε τι λεπτομέρειε το τι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε μια συμφωνία αεροπορικών μεταφορών. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προωθήσει η Κομισιόν. Εδώ έχουμε ένα πλαίσιο για τους δικούς μας εισηγητές όταν εξετάζουν κάποια συμφωνία που έχει επιτευχθεί και που υποβάλλει η Κομισιόν. Είναι το πλαίσιο, επαναλαμβάνω, βάσει του οποίου θα μπορούμε να κρίνουμε κατά πόσον συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Σας το λέω αυτό εισαγωγικά, γιατί οι τρεις τροπολογίες που δεν μπορώ να δεχθώ είναι πολύ λεπτομερείς και πολύ εξαναγκαστικές και δεν είναι γενική και στις κατευθύνες γραμμές. Δεν είμαι δηλαδή για λόγους αρχής εναντίον τους ή θεωρώ ότι είναι εσφαλμένες τροπολογίες. Όχι, καθόλου. Απλώς θεωρώ ότι δεν έχουν θέση σε αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό. Μπορούμε να εξάσουμε ίσως κάποιες από τις τροπολογίες. Τροπολογία 1, Runner, που να φέρει ρητά το τι έχει αναλάβει σαν δέσμευση η Επιτροπή, να σέβει την αρχή τη σχέση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Προφανώ αυτό το υποστηρίζουμε. Υπάρχει η τραπολογία 9 τη κυρία Δεβεράκ που αναφέρεται στην αρχή τη ισορροπή προσέγγιση όπω αυτή βρίσκεται στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτική Αεροπορία και αυτό νομίζω είναι πολύ σωστό. Και επίση μπορώ κάλλιστα να υποστηρίξω τι τροπολογίε τη κυρία Μάισνερ που ζητά όλους, όλα τα κύρια μέρη μια συμφωνίας να συμφωνήσουμε με τι διατάξει που έχουν οριστεί. Επίσης, τροπολογία 4 που καλύπτει το θέμα της υπερπτωσής τη Ιβυρία. Και ακριβώς αυτό το θέμα, αυτή είναι μία από τις προφορικές απολογίες τις οποίες θέλω να με τη 10 και την 11 έχω προβλήματα που αναφέρει την εισαγωγή νομοθεσίας για την προστασία της υγείας του πληρώματος. Παναλαμβάνω ότι είναι πολύ περιουσιαστικό, Όχι ότι είμαι αντίθετη με το θέμα της προστασίας του πληρώματος ή της πρόβλεψης ζωνών ασφαλείας για τα παιδιά κάτω των δύο ετών, αλλά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό το θέμα μέτρων ασφαλείας στα αεροσκάφη. Προσπάθησα να καλύψω τα γενικά θέματα ασφαλείας σε άλλες παραγράφους χωρίς να είμαι τόσο, τόσο λεπτομερής. Όταν υπάρχουν λοιπόν διαπραγματεύσει με τρίτες χώρες υπάρχουν ήδη οι κανονισμοί ασφάλειας. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 15 της κυρίας Ράνερ δεν θέλω να την υποστηρίξω γιατί δεν νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ισορροπήσουμε το θέμα των ισχυρών και αδυνάτων σημείων των ισχυρών συμφωνιών. Δεν διαφορώ με την αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη μέθοδος. Αυτό σας θα πρέπει να το εξετάσουμε στο μέλλον, να δούμε πώς θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, το παραδέχομαι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό εδώ που προτείνεται είναι η καλύτερη άγουσα για να πετύχουμε αυτή την γενική εικόνα. Γι' αυτό έχω βάλει μείον σε αυτή την τροπολογία 15, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος και δεν θα ήθελα να μπει τίποτα στην ε, έκθεση με το οποίο να μην μπορώ να συμφωνήσω. Αυτή είναι οι απόψη μου και θα ήθελα να ξανατονίσω. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί συναδελφοί, ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο, κατευθύντρια γραμμή που οποία θα πρέπει να εργαστούν οι βουλευτέ όταν πρόκειται να αξιολογήσουν μια συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με μια τρίτη χώρα, τρίτο συμβαλόμενο μέρο. Δεν είναι μια συγκεκριμένο κανονισμό που ελέγχει την αερομεταφορική βιομηχανία του των λεχθένων, η κυρία Ράνερ έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ευχαριστώ τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή έκθεσή του. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην έκθεση αυτή υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει στο μέλλον το Κοινοβούλιο μια νομική κατάσταση. Από όσα μας είπατε, πραγματικά συμφωνούμε πρόκειται για ε, συμφωνίες πλαίσιο που ορίζουν γενικές κατευθύνες γραμμές, αλλά δεν θα πρέπει να μπούμε στις λεπτομέρειες. Καταρχήν δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι λεπτομέρειες και ε, επίσης αυτό θα εξαρτάται από κάθε συγκεκριμένη συμφωνία. Το ότι θα πρέπει δηλαδή να ληφθεί εκάστοτε ιδιαίτερη υπόψη. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ειδικέ κατευθυντήρε γραμμέ, όπω προτείνετε και εσεί. όσον αφορά την άποψη ε, για την τροπολογία μου 15, έχω να προσθέσω ότι θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την εργασία μας στο Κοινοβούλιο και στις πολιτικές ομάδες, αν στο μέλλον η Κομισιόν μας έλεγε ποια είναι τα δύνατα και τα δυνατά σημεία μιας συμφωνίας. γιατί συνήθως μας στέλνουν μια τέτοια συμφωνία, πρέπει να τη συζητήσουμε, να αποφασίσουμε υπέρ ή κατά χωρίς όμως να ξέρουμε πού υπάρχουν ενδεχομένω προβλήματα. Θα ήταν καλύτερο λοιπόν να μας ενημέρωνε η Κομισιόν με ποιες από τις διατάξεις της συμφωνίας έχουμε καλές εμπειρίες από το παρελθόν, με ποιες όχι. Ε, αυτό θα ήταν ένα πλεονέκτημα. Ε, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο μόνο τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που θα θέλω είναι να μας δίνει η Κομισιόν μετά διαπραγματεύσει των συμφωνιών περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σημεία, συμφωνούμε απόλυτα νομίζω. Ευχαριστώ. Ο κ. Αλκαντράουι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Η έκθεση καλύπτει όλα τα σημαντικά σημεία, της διεθνής ε, μεταφορές για τις αεροπορικές εταιρείες. Ζητάτε επίσης ε, πιο ανοιχτό και ολοκληρωμένο ε, σύστημα και αγορά αεροπορικών μεταφορών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει να λυθεί υπόψη η ασφάλεια, η περιβαλλοντική προστασία, όλα τα θέματα. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε την επίπτωση αυτών των συμφωνιών και στους εργαζόμενους από την ε, θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο και τα κυβουλευτές έχουν περισσότερες ε, αρμοδιότητες. Θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Η ομάδα μου θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να οργανωθούμε τα επόμενα χρόνια, να δούμε ποια προσέγγιση θα έχουμε, τι ρόλο θα παίξει η Κομισιόν στις στη δουλειά μας. Έχουν δημιουργηθεί διάφοροι νέοι φορείς. Έχουμε αυτές τις κοινέ ας επιτροπές, οι οποίες θα εμπλακούν στην, ε, στις ρυθμίσεις και, στην, και στις αδειοδοτήσεις. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή μας να γνωρίζει τι κάνουν όλοι αυτοί οι φορείς. Επίσης συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς τις τροπολογίες. Οι περισσότερες είναι πολύ καλές και στις περισσότερες περιπτώσεις εξασφαλίζουν ένα πιο έντονο και συγκεκριμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με τον συντάκτη ότι δεν θα πρέπει, και με την κυρία Λίχτεμπεργκ, ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε σε λεπτομέρειες. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο mm. κάποια σημεία την αξιολόγηση Πώ θα το εκφράσουμε δηλαδή, το σημείο αυτό καλύτερα. Αλλιώ ε, ε, μπορεί μετά από λίγα χρόνια να θέσουμε τα ίδια ερωτήματα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων αυτών των συμφωνιών. Αν δηλαδή έχουν επιτύχει τους στόχους τους, ε, αν έχουν πετύχει αυτά που υποσχέθηκαν κτλ. Αξίζει να κοιτάξουμε προηγούμενες συμφωνίες για να δούμε αν οι αρχικοί στόχοι υλοποιήθηκαν ε, μετά από αξιολόγηση μετά από κάποια χρόνια. Φυσικά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε... Κυρία Μάσνερ, σας ευχαριστώ. Ε, ακούσαμε πολλά εγωδιαστικά λόγια και δεν μπορώ να συμφωνήσω. Όλα τα είχατε κανονό. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπίσουμε τα συμφέροντά μας που αφορούν τις ε, συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ορισμένα πράγματα όπως παραδείγματος δίκαιο ανταγωνισμού, αποφυγή επικαλύψεων, ανταλλαγή στοιχείων αλλά και προστασία στοιχείων. Όλα αυτά εδώ συμπεριλαμβάνουν και ταυτόχρονα θα μπορούσα να είμαι σύντομη και να περάσω αμέσω σε λόγο τροπολογίες. Έχω εδώ την τροπολογία μου 3 για να διευκρινίσω ότι δεν λείπει μόνο η Ινδία και η Κίνα, αλλά και η Ιαπωνία και η Ρωσία. Και αυτό για μας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να καλύψουμε και τις μεγάλες αυτές ε, ε, χώρες. Είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε και με αυτές κάποιες συμφωνίες. Κύριε Σιγητά, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας όσον αφορά την αξιολόγηση των τροπολογίες. γιατί πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι οι 10 και η 11 που είναι πάρα πολύ σημαντική και όσον αφορά την ασφάλεια του πληρώματος αλλά και την ασφάλεια των παιδιών, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά αυτό δεν ε, ταιριάζει βέβαια να μπει εδώ στην ε, ε, έκθεση αυτή για τον κανονισμό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά μέτρα για την ασφαλή των παιδιών και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθούν εδώ σε αυτή τη συμφωνία πλαίσια. Εκεί που διαφωνώ με τον Brian Simpson είναι η τροπολογία 15. Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε κάθε πληροφορία, κάθε στιγμή από την Κομισιόν. Και γι' αυτό η δική μου ομάδα, η άλλη, είναι υπέρ του σημείου 15 και θέλω να πούμε ότι κάθε στιγμή χρειαζόμαστε τις πληροφορίες. Και η Κομισιόν θα μπορούσε οπωσδήποτε και να μας τις δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή που είναι ε, αρκετά καλή και και σας ευχαριστώ και για τις ε, ε, που αφορούν τις ε, εκπομπές ε, που έχουν σημασία για τις κλαματικές αλλαγές. Τώρα θα σας πω γιατί αυτές οι δύο τροπολογίες 10 και 11 έχουν υποβληθεί από μένα γιατί ακριβώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ασκήσουμε κάποια άλλη, κάπου αλλού μάλλον επίδραση. Δεν έχουμε κάποιο φάκελο σχετικό, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αναφερθεί εδώ μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα πάντα τα δοκιμάσαμε και αυτό προσπάθησα εδώ να υπενθυμίσω ότι δεν πρόκειται μόνο για χρήματα και ανταγωνισμό και αγορές ε, αεροπορικών επιχειρήσεων κλπ. Αλλά ότι οι αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να είναι ασφαλείς για εκείνους που συνεχώς πετάνε το πλήρωνα δηλαδή και το ειδικό θέμα που μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα των καθισμάτων για τα παιδιά. Γι' αυτό το συμπεριέλαβα. Γιατί αλλού δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε οτιδήποτε. ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Απορρίπτονται τα πάντα, καταπολεμούνται τα πάντα. Άλλο σημείο. Θα ήθελα να υποστηρίξω και την ε, τροπολογία 15 της κυρίας ε, Ράνερ, γιατί και στο SWIFT και στις, ε, στην αρχή των διαπραγματεύσεων PNR είδαμε τι γίνεται, ότι οι πληροφορίες από πλευράς Κομισιών είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται συνεχώς και με πληρότητα. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναφερόμαστε σε θέματα αρχής ε, πολύ γενικά Παρά άμα εξτάζουμε μια συγκεκριμένη ε, συμφωνία, λέμε δεν ταιριάζει αυτό, δεν ταιριάζει εκείνο, δεν ταιριάζει το άλλο. Ταιριάζει μονάχα εκείνο που είναι προ όφελο των μεγάλων ανταγωνιστών. Σε αεροπορικέ μεταφορέ έχουμε δύσκολη κατάσταση. Να προσπίσουμε τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, των εργαζομένων. Γιατί ακριβώς από την άλλη μεριά είναι τόσο έντονη η ισχύς της άλλης πλευράς, όπως είπαμε. Και γι' αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου κακή ιδέα το να υπάρχει η ανάγκη υποβολής των στοιχείων αυτών, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε ουσιαστικά θέματα. Το έβρος των φωνών, τη τηρησή κλπ. Και αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω και εγώ την τροπολογία αυτή. Κατά τα άλλα, οτιδήποτε οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια και οτιδήποτε συμβάλλει στο να μην αποκλειστεί το Κοινοβούλιο σε τέτοια θέματα, μπορώ απόλυτα να το υποστηρίξω μέσα στα πλαίσια της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια από τα θέματα που θέσατε και εσείς θέλω να θέσω και εγώ. Ε, οι τροπολογίες, πολλές από τις τροπολογίες είναι συγκληρωματικές ε, με το αρχικό σας κείμενο. Κάποιες όμως ε, της κυρίας Ράνερ και της κυρίας Λίχτεμπερ ξεπερνούν ε, το αντικείμενό μας. Εδώ, όπως είπατε, πρέπει να είναι ευρείες κατευθυντήριες γραμμές, ενδεδειγμένες, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ενώ αυτές οι τροπολογίες μπαίνουν σε τέτοιες λεπτομέρειες. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε αυτή τη θέση, ε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες. Εμπλεκόμαστε περισσότερο στα τεκτενόμενα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτές οι συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες αντικαθιστούν κυρίως διμερείς συμφωνίες που ήταν ενισχύει επί δεκαετίες με τρίτες χώρες. Το να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εμπιστευόμαστε την ε, Κομισιόν και λέμε όμως ότι επανερχόμαστε στις συμφωνίες αυτό, αυτές και τις ξαναελέγχουμε, θα ήταν μη ρεαλιστικό και δύσκολο. Ανησυχώ επίσης για τα κοινωνικά θέματα. Το να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες συμφωνίες δηλαδή για να ε, επι, ε, επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ε, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ημών και, και των ΗΠΑ. Ε, είμαστε αρκετά επιθετικοί για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η άποψή, μας, ε, η άποψή μου δεν έχει αλλάξει. Η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει, λέει, ότι εμπλεκόμαστε στη διαδικασία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς η Επιτροπή μα ή το κοινοβούλιο. Δεν είμαστε διαπραγματεύσει. Η Κομισιόν η διαπραγματεύτρια. Και γενικά δεν κάνει άσχημη δουλειά. Και σωστά υπόθηκε αυτό που υπόθηκε, ότι οι συμφωνίες αυτές ε, ε, με την Κίνα, ας πούμε, ή με άλλες ευαίσθητες χώρες, με μεγάλους εμπορικούς εταίρους, είναι πολύ σημαντικές. Ε, το τελικό μου σχόλιο τώρα είναι ότι κάποιες από αυτές οι αποφάσεις για διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών είναι στρατηγική σημασία και θα είναι δύσκολο η, Κομισιόν να μας βρει όλους σύμφωνους. σας εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω να μας ενημερώνετε, να μας δίνετε τις πληροφορίες που θα χρειαστούμε. Ακούστε τις, τα σχόλια που θα κάνει η Επιτροπή μας, ε, που θα είναι και σημαντικά σε ορισμένε περιπτώσεις. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε μαζί να υποβάλουμε μια προφορική τροπολογία. Ζητώντας από την Επιτροπή οποιοδήποτε είδους διαπραγματεύσεις για τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας εκεί πάντοτε ρητός να αναφέρεται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο και να ζητείται γνώμη του σε σχέση με οποιαδήποτε ύστερη τροποποίηση των διεθνών συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και τρίτων χωρών. Υπάρχει μια διαδικασία για την τροποποίηση των συμφωνιών αυτών. Είναι σημαντικό ωστόσο να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε σε σχέση με τέτοιες μελλοντικέ τροποποίησεις και πρέπει να αναφέρεται ρητό στο κείμενο της συμφωνίας ότι για οποιαδήποτε ύστερη τροποποίηση ενημερώνεται το κοινοβούλιο και ζητεί τη γνώμη του. Ευχαριστώ. Κυρία Γέγκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ Καταρχά εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να πω ότι καλωσορίζουμε την έκθεσή σα. Βλέπουμε ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και αυτό είναι βάση ε, των εργασιών μας για οποιαδήποτε μελλοντική διεθνή συμφωνία. Να υπεγραμμίσω επίσης ότι συμφωνούμε με την έκθεση. Εν γέννη συμφωνούμε και με τα σχόλια που κάνατε για τι τροπολογίε. Πιστεύουμε ότι κάποιες είναι υπερπεριοριστικές, για κάποιες χρειαζόμαστε ειδική εντολή, κάποιες υπερβαίνουν το πλαίσιο των, ε, των συμφωνιών, πάντως εκτιμούμε τη δουλειά που κάνατε. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να επανεπιβεβαιώσω εκ μέρους ε, του Αντιπροέδρου Κάλλας και της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης τη βούλησή μας ε, να τηρούμε πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις μελλοντικές εξελίξεις. Θα συμφωνήσετε επίσης μαζί μου ότι οι διεθνεί διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές ως προς το χαρακτήρα τους, μεταβάλλονται τάχιστα, ιδίως ε, όταν πλησιάζει η ολοκλήρωσή τους. Και κατά το παρελθόν πάντοτε μας, σας ενημερώναμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως παραδείγματο χάρη την τελευταία φορά όταν κάναμε τις διαπραγματεύσεις μας στην Καμπέρα για τη Και σας είπαμε ότι θα ενημερώνεστε πλήρως για όλες τις εξελίξεις. Θα υπάρχει ε, συγγνώμη, και κλεισμένο των θύρων είχαν γίνει αυτέ οι ε, διαπραγματεύσει. Πάντοτε όμω θα σα τηρούμε ενήμερου. Το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον. Βέβαια, υπάρχει και ζήτημα εμπιστευτικότητα. Να δούμε και τα θέματα διαφάνεια όμω. Ελπίζω να καταφέρουμε να συμφιλειώσουμε αυτά τα δύο. Θέλω να σα ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την έκθεσή σα, κύριε Πρόεδρε. Και ολοκληρώνοντα, εκφράζω εκ νέου την πλήρη δέσμευση και την ε, επιθυμία της Κομισιόν να συνεργαστεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια σημεία. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου αλλά και τις υποχρεώσεις του, εγώ πιστεύω ότι ε, αν δείτε την έκθεση και αν δείτε συγκεκριμένα τις παραγράφους 12, 13, 14, στην παράγραφο 12 λέγεται ότι για να μπορούν να ληφθούν αποφάσει για το κατά πόσο θα δίνεται σύμφωνη γνώμη στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τη διαδικασία από, τις αρχής, θεω, από την αρχή. Συγγνώμη, θεωρεί ότι είναι επίση προ το συμφέρον των άλλων θεσμικών οργάνων τυχώ ανησυχίε ιδιαίτερη σημασία που θέτουν που αμφισβήτη στην θεμότητα του Κοινοβουλίου να παράσχει την έγκρισή του, να εντοπίζονται και να καθησυχάζονται σε αρχικό στάδιο. Πέν ότι η Συμφωνία Πλαίσιο 2005 δεσμεύει ήδη την Επιτροπή να παρέχει έγκαιρη και σαφή ενημέρωση στο Κοινοβούλιο κατά την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση των διεθνών διαπραγματεύσεων. Πόσο πιο ξεκάθαρα να τα πω σε σχέση με τις υποχρεώσεις. Και μετά λέει, αναμένει από την, επιτροχή, την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια Επιτροπή, τη δική μας δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση να προταθούν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορέ, τα σχέδια οδηγών διαπραγμάτευσης, σχέδια κειμένων διαπραγμάτευσης και το έγγραφο προς μονογραφή μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες. Τι άλλο να πω στην Επιτροπή, να τους πω μήπως δεν σας εμπιστευόμαστε, την Ευρωπαϊκή Ενώ. Όλα τα άλλα τα έχω γράψει, τα έχω πει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δύο τροπολογίες ε, της Εύα Λίχτενμπέργκερ για τις παιδικές ζώνες τα λοιπά. Εγώ πιστεύω το εξής. Δεν είμαι κατά οποιασδήποτε σχετικής εκστρατείας και συμφωνώ, μαζί σας είμαι. Αλλά δεν είναι αυτό το κατάλληλο κείμενο. Εδώ μιλάμε για διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών αν λέμε ότι θα πρέπει κάτι να γίνει για την ασφάλεια ε, στα αεροσκάφη όταν υπάρχουν μικρά παιδιά μέσα. Ναι, συμφωνώ, αλλά όχι εδώ, όχι σε αυτό το κείμενο. Αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει και από πλευράς κρατών μελών σε σχέση με τις διαδεργασίες στο πλαίσιο του, της ΔΟΠΑ. Επίσης, εμείς ξέρουμε ότι έχουμε τις διάφορες ε, οδηγίες όψη οι οποίες ρυθμίζουν τα πράγματα. Όταν μιλάμε για τρίτες χώρες και αν θέλουμε να ασκήσουμε πιέσεις, ναι, θέλουμε να είναι ασφαλείς μεταφορές. Και κάπου στην έκθεση τα λέω αυτά. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει εποπτεία, έλεγχος για τον τομέα της ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό καλύπτεται. Είναι περιοριστικές τροπολογίες, εντάξει δεν μπορώ να επιμείνω πάντοτε θα σέβομαι την άποψη των περισσότερων μελών της Επιτροπής μας και θα δούμε τι θα γίνει αύριο και στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάντως όλες και όλους για τη συνεισφορά σας και θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Μην ξεχνάτε όμως ότι εδώ μιλάμε για ένα πλαίσιο που πρέπει να συγκροτεί η Επιτροπή και εντό του οποίου πλαίσιο πρέπει να εργάζονται και στο μέλλον όλοι οι συγητές και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Πάμε στους ελκυστήρες τώρα. Από τα Α380. Λοιπόν, η κυρία Σεναλόβα θα μας μιλήσει για τις διατάξεις που αφορούν τους κινητήρες που διατίθεται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος για τους ελκυστήρες. Αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΝΒΗ θα ψηφίσουν αυτήν την εβδομάδα. Κυρία Σεναλόβα, έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή η έκθεση συνδέεται με την οδηγία που υιοθετήσαμε πριν από δύο μήνες και όπως είπατε κι εσείς, η υπεύθυνη. Επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΜΒΗ. Εκεί θα γίνει η ουσιαστική συζήτηση, η βασική συζήτηση για την υιοθέτηση ή όχι της έκθεσης. Ποια είναι θέση μου τώρα. Είμαι υπέρ της υιοθέτηση αυτής της έκθεσης, ιδίω σε ό,τι αφορά την επικουρία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προς τον γεωργικό τομέα, αλλά δεν πρέπει να το παρακάνουμε και να πάμε πολύ μακριά ε, στην έκθεση αυτή. Η τροπολογία 1 και 3 είναι τροπολογίες οι οποίες είναι η μία αντιφατική με την άλλη και τελικά δεν υποστηρίζει ούτε τη μία ούτε την άλλη. Η πρώτη ζητάει την ανάκληση της έκθεσης, ενώ η τρίτη ζητάει αντίθετα μία αύξηση της μεταβατικής περίοδου κατά δύο χρόνια. Εγώ ως εισηγήτρια δεν είμαι υπέρ. Αλλά καταλαβαίνω βεβαίως τις α, μεμονωμένες απόψεις. Οι τρεις άλλες τροπολογίες αφορούν διατυπώσεις πιο συγκεκριμένες, ζητούν δηλαδή πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις, δεν έχω πρόβλημα, τις υποστηρίζω και ως εισηγήτρια συνιστώ την υιοθέτηση αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές. Yes. Ευχαριστώ πρόεδρε και μα τι συζητήσεις. δυστυχώ δεν ακόμα έχει έρθει. Γι' αυτό ήθελα να σα πω ότι χαιρετίζω την πρόταση τη ηγετρία. Δυστυχώ δεν μπορούμε να στηρίξουμε την τροπολογία υπερθμών 1, κυρία Λιχτεμπέργερ, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι πάρα πολύ λεπτή η συζήτηση όταν προσπαθούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι κλπ. Θεωρώ ότι η πρόταση της εισηγήτριας στο σύνολό της είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακόμα και η παράταση που ζητάει η κυρία Τίκαο δεν μας φαίνεται ιδιαίτερα προβληματική. Μπορούμε λοιπόν αύριο να υποστηρίξουμε ευρέω την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπέργα. Όχι. Η κυρία Μάσινα πρώτα. Δεν είχα ζητήσει το λόγο ίσω να εγώ φταίω. Δεν ήθελα βέβαια να με παραβλέψετε. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα βέβαια. Γιατί και εδώ, όπως και η έκθεση, ε, μπορώ να συμφωνήσω, κυρία Συνάλλοβα, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έχουμε δύο ε, εκθέσεις. Τέλος πάντων, Το να απορρίψουμε πλήρως και για μένα δεν θα ήταν η σωστή άγουσα. Γιατί οι λίγες, λίγες ε, μόνο εταιρείε αφορούνται από τους ε, ε, κινητήρες αυτός. Μπορώ λοιπόν να συμφωνήσω. 2013 νομίζω αρκεί. Χρειαζόμαστε ακόμα δύο χρόνια αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρχει και μια νέα οδηγία. Να μην βάλουμε λοιπόν 2013, 2015, ε, συγγνώμη, 2013 αρκεί. Μπορώ λοιπόν απόλυτα να συμφωνήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Η ε, κυρία Λίχτενμπεργκ. Και ε, βέβαια διαφωνώ εδώ. Γιατί νομίζω ότι άμα αποστείλουμε ένα μήνυμα τόσο ήπιο που δεν είναι δυνατή η πραγματική προστασία του κλίματος και μετά προβλέπουμε ακόμα μια αναβολή και ακόμα πιο ελαφρά μέτρα, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ προβληματικό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εάν μέσα στο πλαίσιο του επιχειρήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και θέλουν γι' αυτό να αγνοήσουν το θέμα της προστασίας του κλίματος. Και κάνουν ό,τι μπορούν το σώσουν κατά το δυνατόν αργότερα, πολύ λίγο και ίσως και καθόλου να υιοθετηθούν μέτρα για την προστασία του κλίματος. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω στις κύριου συναδέλφου που και αυτή την Επιτροπή προσπίζουν την προστασία του κλίματος, να τους πω σας παρακαλώ σκεφτείτε το, εάν θέλουμε σοβαρά να αλλάξουμε τη διαδικασία όσον αφορά την προστασία του κλίματος, ορίζοντας κάποιους στόχους εκπομπός, δεν μπορούμε τώρα βήμα προς βήμα Όλου ο ο φακέλος, ο οποίος ίσως είχαμε δείξει και κάποια φιλόδοξη στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναβάλουμε, λέω, όλα αυτά τα θέματα ή τα αποδυναμώσουμε τους φακέλους. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να μείνουμε σοβαροί, θα πρέπει να μπορούν τα θέματα να μείνουν ε, μέσα σε ένα πλαίσιο προβλεπόμενο. Αυτή είναι η δική μου δυσκολία. Τώρα έχουμε ένα φάκελο εδώ που δεν είναι και τόσο σημαντικό όσον αφορά το μέγεθος του τομέα. Εάν το δούνε όμως οι άλλοι θα έρθουν και θα προσπαθήσουν να αποδυναμώσουν όλα τα κριτήρια ξανά και ξανά. Εμείς δεν είμαστε εδώ επιτροπή για την προάσπιση μόνο οικονομικών συμφερόντων. Θα πρέπει να προσπίσουμε και σφαιρικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών. Ίσως κάποιοι μπορέσουν να σκεφτούν κατά πόσον το να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ιδέα, ιδίω μετά τις πρόσφατες καταστροφές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Πεσίν είναι εδώ από την Κομισιόν. Όχι. Η κυρία Σέναλόβα, μήπως θέλει κάτι να προσθέσει. Με όλο το σεβασμό βέβαια. Στον κύριο Ποσινήσης που οπωσδήποτε θα είχε να μας πει πάρα πολύ αξιόλογα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν θα άλλαζαν πολλά τα πράγματα. Η κυρία Σελανόβα όμως, αν θέλει κάτι να προσθέσει, παρακαλώ. No. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε αύριο. Ε, σας παρακαλώ, ε, σταματήστε τον κύριο Βοσελίνη, να μην φύγει. Αύριο ψηφίζουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο είναι η συνεδρία των συντονιστών που θα, θα ξεκινήσει όμως στις 5 και 4 μετά από μία ώρα. Ο Ρόμπερτ δεν είναι εδώ. Ε, δεν ξέρω τι να κάνουμε, να περάσουμε αμέσως ε, στη συνεδρία των συντονιστών. Ε, ο Ρόμπερτ δεν ξέρω, είναι εδώ, νομίζω ότι θα, θα επιστρέψει. Θα σταματήσουμε για πέντε λεπτά και μετά θα αρχίσει ε, η συνεδρία των συντονιστών.